Μάλιστα. Να συνεχιστεί λοιπόν η συνεδρίαση της ομάδας ε, που ξεκίνησε σήμερα το πρωί. Σας παρακαλώ για σταματήστε τις συζητήσεις για να δώσουμε την απαραίτητη πρόσοχη εδώ στην αίθουσα να σας υποδείξω εκ νέου ότι η συνεδρίαση ε, μεταδίδεται στο διαδίκτυο έχουμε μαζί μας και μία σειρά δημοσιογράφων. Να καλωσορίσω λοιπόν καταρχάς εκ βάθους καρδίας τον Ζαν Κλόντ Ιούγκερ, ο οποίος είναι υποψήφιος ε, και ως τέτοιος υποψήφιος ε, θα ε, ψηφιστεί για τη θέση του θέλει να ψηφιστεί για τη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Τον καλέσαμε λοιπόν τον Ζαν Κλόντ Ιούγκερ γιατί θεωρώ ότι αυτό ε, είναι τμήμα της δημοκρατικής κουλτούρας ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, της ομάδας μου. Το ίδιο κάναμε πριν από πέντε χρόνια και με τον κύριο Μπαρός. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που κάναμε τότε. Θα ήθελα εν συντομία να παρουσιάσω τον κύριο Γιούνκερ στην ομάδα, αν και είμαι βέβαιη ότι γνωρίζετε τον κύριο Γιούγκερ και γνωρίζει και ο ίδιος σε ποια ομάδα βρίσκεται. Η ομάδα αυξήθηκε αριθμητικά στις ευρωεκλογέ 52 μέλη και είμαστε σε αντίθεση με τις άλλες ομάδες μια ομάδα ομοσπονδιακή. Δηλαδή, η πολιτική ομάδα αποδέχεται την ε, πολυμορφία της και τη διαφορετικότητα των μελών της. Και θεωρώ ότι αυτό είναι εξαιρετικό για το ευρωπαϊκό συγκείμενο την ποικιλομορφία των σοσιαλιστικών ε, αριστερών, κομμουνιστικών ε, δυνάμεων και συνιστώσεων. Η δύναμή μας λοιπόν είναι στην πολυμορφία μας. Και γι' αυτό λοιπόν αν υπομονώ πραγματικά να ακούσω και τις ερωτήσει ε, που θα σας τεθούν σήμερα κύριε Γιούγκερ. Συμφωνήσαμε ε, επί της εξής μεθόδου, την οποία και έχω ήδη παρουσιάσει στα μέλη. Έχουμε 19 αντιπροσωπείες εδώ στην ομάδα, 19 κάθε αντιπροσωπεία ανεξάρτητα από τα αριθμητικά της, από την αριθματική της δύναμη έχει τα ίδια δικαιώματα. Εσείς λοιπόν έχετε 10 έως 15 λεπτά στη διάθεσή σας για να μας πείτε πώς σκοπεύετε να επιτελέσετε το έργο σας αν εκλεγείτε ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς ε, ενδιαφερόμαστε φυσικά ιδιαιτέρως για θέματα του πώς θέλετε να αλλάξετε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στην Τρόικα, στην ε, εφαρμογή των δραστικών πολιτικών ε, λιτότητας και περικοπής, περικοπών, το πώς μπορεί να ενισχυθεί η αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πώς θεωρείται ότι η ψήφος εκατομμυρίων ψηφοφόρων μπορεί να ερμηνευθεί και να εφαρμοστεί ποιες θα είναι οι δικές σας αντιδράσεις αυτή την σαφή κριτική που ασκήθηκε για την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα και τέλος πώς μπορεί να γίνουν σημαντικές διορθώσεις. Τι θα κάνουμε λοιπόν όταν θα λάβατε το λόγο και θα έχετε ολοκληρώσει την εισαγωγή σας, θα πάρουν το λόγο η επικεφαλής των αντιπροσωπιών ή όποιος θέλει από την κάθε αντιπροσωπεία έως δύο λεπτά. Επιμένω σε αυτό. Και μετά από πέντε ομιλητές θα σας δίνω το λόγο για να απαντήσετε. Συμφωνείτε? Περνάμε λοιπόν κατευθείαν στην εισαγωγή, ξεκινάτε και έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Με ιδιαίτερη χαρά ανταποκρίθηκα στην πρόκληση της πολυφωνικής αριστεράς, αν μου επιτραπεί η έκφραση. Ε, γνωρίζω καλά την ομάδα σας, διότι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή και λιγότερο ενίοτε παρακολούθησα ε, τις εργασίες σας καθώς ε, και τις προεκλογικές εκστρατείες όλων όσων παρευρίσκονται ε, στην σημερινή συνεδρία. Σε σχέση τώρα με την έκβαση των συζητήσεων μας, ε, δεν έχω καμία αμφιβολία. Ο κύριος ε, Μελανσό με έχει ήδη απειλήσει ότι μου έχει διάφορα φυλαγμένα, οπότε καταλαβαίνω ότι θα είναι δύσκολη η έκβαση των ε, συζητήσεων, αλλά δεν με εντυπωσιάζει αυτό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών. Δεν θέλω να μιλήσω για την ιδέα του Σπίτσεν candidate. Ε, υπάρχουν αυτοί που είναι υπέρ, ε, κατά και Πιστεύω ότι στα πλαίσια της άμεσης καθολικής ψηφοφορίας είχε αυτό νόημα και την επόμενη φορά πιστεύω ότι αυτό το επιπρόσθετο δημοκρατικό στοιχείο θα επιτρέψει ε, στους ευρωβουλευτές να έχουν έναν ενισχυμένο ρόλο την επόμενη δεκαετία σε σχέση με τις προηγούμενες. Λοιπόν, τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών ε, με οδηγούν σε διάφορες σκέψεις, όπως και άλλοι, αλλά δεν σημαίνει αυτό ε, τίποτα. Διαπιστώνω ότι υπάρχει ένα διευρυνόμενο χάσμα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες της. Αυτό οφείλεται στην Ευρώπη σε κακές πολιτικές, ατελείς ε, πολιτικές ε, σε εθνικά ε, αντανακλαστικά που βλέπουμε σε επίπεδο κυβερνήσεων αλλά και σε επίπεδο διεθνούς κοινή γνώμης. Οι πολιτικοί ηθήνοντες που καταλαμβάνουν διεθνή αξιώματα όπως εγώ στο παρελθόν και ελπίζω και στο μέλλον είναι σε θέση να καταλάβουν τα τεκτενόμενα στην Ευρώπη και εύκολα μπορεί κάποιο σε εθνικό επίπεδο να καταγγείλει ε, τις ε, αποφάσεις που από κοινού όμως ελήφθησαν ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τελικά προκαλείται μια μεγάλη σύγχυση. Υπάρχουν κάποιοι που δεν αγαπούν, που δεν θέλουν την Ευρώπη από αυτού που ψήφισαν, που είναι ρατσιστέ, μυσαλόδοξοι, ε, που ε, αγαπούν μόνο τους εαυτούς τους, ε, για του οποίου, το χρώμα του δέρματο, ο σεξουαλικό προσανατολισμό, οι φιλοσοφικές πεπιθήσεις αποτελούν στοιχεία απόρριψης ε, του εταίρου ε, και έχουμε ακροδεξιά, ε, σκληρή ακροδεξιά και αν εκλεγώ δεν θα υπάρξει κανένας διάλογος μαζί τους. Δεν πρόκειται να ξεκινήσω κανέναν διάλογο με τους εκπροσώπους αυτής της λυπηρής εκτροπής της δημοκρατικής ευρωπαϊκής σκέψης. Οι απαντήσεις δεν πρέπει να είναι ούτε υπερβολικά απλωστευμένες ούτε υπερβολικά περίπλοκες. Υπάρχουν ε, πέρα από τους λαϊκιστές ε, κάποιοι που θεωρούν ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο δεν ανταποκρίνεται πλέον στις προσδοκίες τους. Ευελπιστώ να ξεκινήσει ένας ενάρετος κύκλος συζητήσεων με αυτούς τους ανθρώπους που θα οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και δεν σας κρύβω ότι αυτοί που ψήφισαν για τις κλασικές μεγάλες ευρωπαϊκές πολιτικές οικογένειες ε, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως απλοϊκοί, ως κάποιοι που δεν έχουν ενστάσεις να προβάλλουν σε σχέση με το ευρωπαϊκό σχέδιο όπως διαμορφώνεται σήμερα. Πιστεύω ότι το πραγματικό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών αυτής ε, είναι, περιστρέφεται μάλλον γύρω από την ανάπτυξη και από την απασχόληση. Ε, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ε, ως προς την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την ενέργεια, τα ταλέντα, τη δυναμική της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα προσιλωθώ σε αυτό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δώσουμε την εντύπωση ότι μπορούμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης. Όχι, ένα γενικό πλαίσιο μπορούμε να στήσουμε ούτως ώστε να αναπτυχθεί ε, η αγορά εργασίας, να δημιουργηθούν οι απαιτούμενες συνθήκες ώστε να έχουμε μια μη πληθωριστική ανάπτυξη και ως εκ να δημιουργηθούν και θέσεις απασχόλησης ε, στην Ευρώπη. Καθόλου σχεδόν ε, την ε, διάρκεια της πολιτικής μου ζωής μπορεί να θεωρείται ότι έχω απλοϊκές ιδέες σε σχέση με την αγορά εργασίας. Όσοι γνωρίζουν τα πιστεύω μου για αυτό το θέμα θα συνειδητοποιούν ήδη ότι βάσει του πολιτικού πολιτικού μου λόγου ποτέ δεν δέχτηκα να ε, βυθιστώ ε, ε, στον κρεμό του νέου φιλελευθερισμού και να προσπαθήσω εκεί να βρω απαντήσεις. Χρειαζόμαστε έναν υγειονομικό κλειό γύρω από ένα, συγγνώμη, ένα δίχτυ ασφαλείας για τις αγορές εργασίας για να αποφύγουμε οποιασδήποτε υπερβολές, οποιασδήποτε παρεκτροπές μπορούν να ανακύψουν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να ξέρουμε και παρότι ότι κάποιοι δεν θέλουν να το λένε, ότι δεν μπορούμε να δαπανίσουμε κονδύλια που δεν έχουμε. Σίγουρα μπορούμε να συλλέξουμε ε, κονδύλια ε, εκεί όπου παλιά ε, τα κράτη-μέλη δεν παρενέβαιναν σε φορολογικό επίπεδο και αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Πιστεύω ότι ως προς την οικονομική ε, και ε, νομισματική πολιτική και το ευρώ και αναφερθήκατε και εσείς στην Τρόικα Είχαμε κάποια καλά αποτελέσματα διότι ε, παρότι ήταν δυσχερέστατο το εγχείρημα καταφέραμε να διατηρήσουμε λοιπόν την Ευρωζώνη ως πρόεδρος αυτής αγωνίστηκα για αυτό το στόχο ε, προσπαθήσαμε και καταφέραμε να ε, καταπολεμήσουμε ε, την τάση αποκλεισμού της Ελλάδας, να διατηρήσουμε μια εσωτερική συνέπεια ακολουθία στην Ευρωζώνη. Είχαμε στη διάθεσή μας όχι ιδανικά εργαλεία, αλλά σίγουρα είχαμε κάποια εργαλεία, γιατί σε άλλες περιπτώσεις δεν υπήρχαν. Έπιασε φωτιά το αεροπλάνο στον αέρα και ξέρετε έπρεπε να αντιδράσουμε άμεσα και δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Για την Τρόικα ε, έχω πολλές σκέψεις που μπορώ να καταθέσω ενώπιον σας. Εγώ ε, στην Ευρωζώνη δεν ήμουν υπέρ της παρέμβασης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στους μηχανισμούς ε, διάσωσης της ευρωπαϊκής οικονομίας και τελικά μου εξήγησαν και αληθεύει αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συνηθίσει να μαγειρεύει τέτοια προγράμματα διότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει την τεχνογνωσία ότι θα έπρεπε να ε, συμμετάσχει σε αυτό το μηχανισμό. Εγώ ε, ανέκαθεν ε, να επικρίσεις στο Διεθνώς Νομισματικό Ταμείο για τις λύσεις που πρότεινε σε διάφορες περιπτώσεις. Είδαμε ότι προχώρησε η συζήτηση με τη Λαγκάρ και το Διεθνές Συγγνώμη Νομισματικό Ταμείο και τελικά μπορούσαμε να βρούμε λύσεις προσαρμοσμένες ε, στα διάφορα προβλήματα. Ε, μπορούν να αποδοθούν παρόλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, κάποια εύσημα ε, στην Τρόικα. Διαπιστώνω εκεί ένα δημοκρατικό έλλειμμα. Δεν καταδικάζω λοιπόν την ίδια την Τρόικα. Θα πρέπει να τροποποιηθεί η φύση της, να καταστεί πιο δημοκρατική και να καλυφθούν τα ελαττώματά της. οι κρατικές αλλά και ιδιωτικές επενδύσεις στην Ευρώπη έχουν γνωρίσει μια θλιβερή μείωση. Η αναπτυξιακή πολιτική φαίνεται να είναι μια παράλληλη πολιτική. Στον επενδυτικό χώρο δεν πρόκειται να μας δώσει ε, κανένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εξετάζουμε τώρα τα ενδεχόμενα, τις δυνατότητες που υπάρχουν, ώστε να τονώσουμε έτσι περαιτέρω την Ευρωπαϊκή Βούληση να αυξήσει ε, τις επενδύσεις, ε, να ενισχύσει τα υφιστάμενα εργαλεία και ενδεχομένως να προσθέσουμε στα ε, εθνικά και ευρωπαϊκά οπλοστάσια νέα χρηματοπιστωτικά εργαλεία πέρα από το υφιστάμενο εργαλείο της αποκατάστασης των χρηματοοικονομικών ροών με αποδέκτες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιθυμώ να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος ε, ως προς την δημοσιονομική ε, σύγκληση, ε, ως προς τη φορολόγηση των επιχειρήσεων θα ήθελα να πω συγκεκριμένα ότι είναι αδιαμφισβήτητη η ανάγκη να συμφωνήσουμε επί κοινών αξώνων ως προς το, τη φορολογική βάση την, ε, για την κοινή ε, φορολογική βάση έχουν γίνει ήδη προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως επίσης έχουν κατατεθεί προτάσεις και για το FTT, για τον ε, φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, που παραμένουν υπό εξέταση από την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Θα πρέπει να είμαστε πιο εμπνευσμένοι και ανέκαθεν συνηγορούσα υπέρ ενός ελαχίστου κοινωνικού μισθού. Με οδηγία δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε αυτό. Σε κανένα κράτος μέλος μπορούμε όμως να φροντίσουμε να υπάρχει ένα, ένα ελάχιστο, ένας ελάχιστος μισθός που θα προβλέπεται σε εθνικό επίπεδο. Οποιοςδήποτε εργάζεται θα πρέπει να μπορεί να ζει από τους καρπούς ε, της εργασίας του και επίσης ε, ε, θα πρέπει να υπάρχουν ίσες αμοιβέ σε περίπτωση απόσπασης αυτός που αποσπάται από κάποια επιχείρηση σε άλλη χώρα φυσικά θα πρέπει να λαμβάνει ίση αμοιβή επί τη βάση ή ε, της νομικής ε, τάξης που ισχύει σε κάθε κράτος μέλος ή βάσει των συμβατικών υποχρεώσεων που ισχύουν ε, σε όλες τις συμβάσεις έχει συνάψει η επιχείρηση. Δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία διαφοροποίηση ως προς τις απολαβές αυτών των εργαζομένων εάν εκλεγώ Πιστεύω ότι θα ε, τονίσω πόσο σημαντικό είναι κανείς να συνδικαλίζεται, ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να ανήκει κανείς σε ένα συνδικάτο από ότι ε, σε μία ε, πολιτική ομάδα. Παρότι ήμουν σε χριστιανοδημοκρατικό συνδικάτο, δεν σημαίνει τίποτα αυτό, ούτε και σημαίνει Ε, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να μετέχει κανείς στο συνδικαλιστικό κίνημα. Τώρα το ε, φορολογικό και το κοινωνικό dumping είναι ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν με μεγαλύτερο ενδιαφέρον από όλους όσους προετοιμάζουν τις πολιτικές αποφάσεις είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε εθνικό επίπεδο. Εγώ θα ήθελα ε, για τη μετανάσταψη, παραδείγματος χάρη να ασχοληθούμε με το σύνομο αλλά και το έκνομο κομμάτι της. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές ε, στα νομικά συστήματα των κρατών μελών και ε, χρειάζονται πολλές διορθωτικές δράσεις ε, σε αυτό το τομέα. Θα ήθελα επίσης να είμαστε ιδιαίτερα φιλόδοξοι ε, για τη συγκρότηση ενός, ε, μιας πραγματικής ενίας ψηφιακής αγοράς, να ολοκληρώνοντας έτσι την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά με τρόπο ώστε η, τα ευρωπαϊκά πρότυπα να μην είναι υποδεέστερα σε σχέση με τους κανόνες της εθνικής αγοράς εργασίας διότι σε κοινωνικό και εθνικό επίπεδο αυτό μας οδηγεί συχνά σε απαράδεκτες καταστάσεις. Στο μέλλον θα ήθελα σε κάποιες χώρες, σε περίπτωση που θα χρειαστεί να υπάρχουν προσαρμογές, αυτό να γίνει με άλλη μεθοδολογία. Περίπτωση που παρουσιαστεί ανάγκη. Ο κοινωνικός αντίκτυπος ε, των ε, μέτρων σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν, θα πρέπει να αξιολογηθούμε με μεγάλη προσοχή και θα ήθελα σε κάθε χώρα τέτοιου προγράμματος σε περίπτωση που υπάρχει τέτοια χώρα και πάλι δεν το καταβάλω αυτό να υπάρχει ένα δεύτερο πλάνο και τα προγνωστικά οι προβλέψεις που αφορούν την ε, οικονομία, την αγορά του εργασίας να μην ε, περιορίζονται σε αυτά που λένε οι διεθνείς εμπειρογνώμονες θα πρέπει να υπάρχει η τάδε ανάπτυξη και αν δεν υπάρχει ανάπτυξη αυτή θα πρέπει να προσαρμόζονται τα προγράμματα σε ό,τι αφορά και την οικονομική κατάσταση και την οικονομική συγκυρία. Αυτό ισχύει για όλο το εύρος των θεμάτων σε ό,τι αφορά το πακέτο σταθερότητα, το σύμφωνο σταθερότητα, ε, όπως και άλλοι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όρισε ότι το σύμφωνο σταθερότητας δεν χρειάζεται αλλαγή. Εγώ το Μάρτιο του 2005 είχα προτείνει μια μεγάλη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας, του πακέτου σταθερότητας που θα μας επέτρεπε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες ευελιξίας που παρέχονται γιατί αυτό χωρίς να υπονομεύσουμε την οικονομική σταθερότητα όλης της Ευρωζώνης αλλά το πακέτο σταθερότητας πρέπει να γίνει με μια μήτρα ανάγνωσης. Και αυτά τα τελευταία χρόνια ε, έχουν αγνοηθεί αρκετά. Και θα έπρεπε λοιπόν να το σκεφτούμε. Νομίζω ότι τα ερωτήματα που θα θέσετε θα έχουν να κάνουν με λεπτομέρειες που θα μας επηρεάσουν. Δεν μίλησα για ευρωπαϊκές αξίες, δεν μίλησα για εξωτερική πολιτική, δεν μίλησα για αμυντική πολιτική, αλλά ήθελα να επικεντρωθώ στην εισαγωγή μου, στις προτεραιότητες εκείνες, οι οποίες θεωρώ ότι είναι οι πιο σημαντικές. Σας ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος, κύριε Γιούγκερ. Και για το γεγονός ότι επικεντρωθήκατε σε κάποια μόνο θέματα. Προφανώς δεν είσαστε εδώ πέρα για να παρουσιάσετε το σύνολο του προγράμματός σας, αλλά χαίρομαι που τα θέματα που αναφέρατε ε, θα είναι και τα θέματα ενδεχομένω στα οποία θα λάβετε ερωτήσεις. Επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, να ξεκινήσουμε κατευθείαν τη συζήτηση και οι διερμηνείς ε, προσφέρθηκαν να μείνουν μέχρι τη μία και τέταρτο περίπου προκειμένου να έχουν την ευκαιρία και οι βουλευτές να απαντηθούν τα ερωτήματά τους. Να ξεκινήσουμε με την Μαρίνα να παρακαλέσω τους συναδέλφους να συστήνονται εν συντομία. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Λέγομαι Μαρίνα Αλβιόλ, είμαι από την Ισκιέρδα Ουνίδα, την ε, Πολυφωνική Ενωτική Αριστερά της Ισπανίας. Κύριε Γιούγκερ, εμείς δεν θα σας στηρίξουμε ως πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και όχι μόνο αυτό, από την πλευρά της ε, η Σκιέρδα Ουνίδα, είμαστε εδώ για να ταχθούμε απέναντί σας και όχι μόνο απέναντί σας, απέναντι σε όλους όσους είστε υπεύθυνοι για τόσο πόνο, τόση οδύνη για να μπορέσετε εσείς οι δικοί σας οι ισχυροί ε, να κερδίζετε εκατομμύρια, ο λαός υποφέρει ε, μέσα στη φτώχεια ε, οι πολιτικές οι οποίες έχουν εφαρμοστεί, οι συντηρητικές πολιτικές σε συνεργασία με τους σοσιαλδημοκράτες και τους φιλελεύθερους επέτρεψαν δισεκατομμύρια κέρδη για τις τράπεζες. Όμως το Ισπανικό κράτος χιλιάδες οικογένειες δεν μπορούν να βάλουν στο τραπέζι ένα πιάτο γεμάτο φαΐ για τα παιδιά τους. Εκατοντάδες οικογένειες ε, αναγκάζονται να υποστούν έξωση από τα σπίτια τους, από τις τράπεζες ή πολλοί νέοι και άλλοι αναγκάζονται να μεταναστεύσουν. Και τι κάνουν οι άνθρωποι που είναι πάνω από 40-50 χρονών και έχουν χάσει τη δουλειά τους χωρίς να έχουν πλέον προοπτικές. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα της πολιτικής λιτότητας που προασπίζεστε εσείς και οι ειδικοί. Επομένως εμείς ποτέ δεν θα γίνουμε συνένοχοι σε αυτή την κατάσταση. Ε, δεν πρόκειται ποτέ ε, να είμαστε στο πλευρό της δεξιάς. Αντίθετα θα την πολεμάμε με όλη μας τη δύναμη. Θα ήθελα πάντως να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις γιατί πολλοί πολίτες μας έχουν ζητήσει να σας θέσουν τα ερωτήματα αυτά γιατί απαιτούν απαντήσεις θα συνεχίσετε να στηρίζετε την Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με τις Ηνωμένε Πολιτείε για την ασφάλεια των τροφίμων, το περιβάλλον, δηλαδή να τα υπαβάλλετε στα συμφέροντα των πολυεθνικών Αμερικανικών εταιριών. Επίσης, τι πιστεύετε κύριε Γιούνκερ για τους φορολογικούς παραδείσους, όπως και το κόμμα σας πιστεύετε ότι στην Θέουτα ή στη Θέουτα η Μελίγια ε, θα συνεχίσουν ε, να υπονομεύονται οι προσπάθειες αυτών που να ζητούν ε, ένα καλύτερο μέλλον. Θα συνεχίσουν ε, οι βομβαρδισμοί στη Γάζα που δολοφονούν αμάχους, αθώους, ε, να μην βρίσκουν μια αντίδραση από εσάς. Και τι έχετε να πείτε για αυτά που γίνονται στην Ισπανία όταν έχουμε δεκάδες εργαζομένων που κινδυνεύουν να μπουν φυλακή επειδή συμμετείχαν σε μαζική απεργία. Δεν είναι δικαίωμα δημοκρατικό αυτό και ολοκληρώνω το Λαϊκό Κόμμα σας στηρίζει και θέλει ε, να αλλάξει το νόμο για την ε, άμβλωση. Να μην μπορούν δηλαδή οι γυναίκες πλέον να αποφασίζουν με ελευθερία γιατί τι θα κάνουν με το σώμα τους και με τη ζωή τους. Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά. Σα ευχαριστώ Μαρίνα Αλμπιόλ, αλλά θα ήθελα να σα υποδείξω το εξή. Έχετε δύο λεπτά μόνο στη διάθεσή σα, Δύο λεπτά. Και σα παρακαλώ μην τα βάζετε όλα τα σημαντικά θέματα σε μία εισήγηση. Θα πρέπει να δείτε τι ερώτηση θέλετε να κάνετε, τι ε, ερωτήσεις έχουν ήδη γενικών, αν και μετά ο κύριος Παπαδημούλης. Σας ευχαριστώ. Είμαι από την ε, Λίνκε. Όσο μιλούσατε, είχα την αίσθηση ότι συνεχίζουν τα πράγματα ως έχουν. Είπατε ότι θέλετε να εκδημοκρατήσετε την Τρόικα και αυτό θέλετε να το αλλάξετε, αλλά γι' αυτό χρειάζεστε και τα άλλα κράτη-μέλη, για παράδειγμα τη Γερμανία. Και δεν ξέρω κατά πόσον θα ήταν ενθουσιασμένη για με τέτοια αλλαγή η Γερμανία. Και αυτό είναι αυτό που σας προσάπτουμε, αυτό είναι που μας ε, κάνει να σας επικρίνουμε. Δύο ερωτήσεις τώρα στη χαμηλή προσέλευση στις ευρωεκλογές βλέπουμε ότι είναι όλο πιο μεγάλο το χάσμα μεταξύ φτωχών και πλουσίων στην Ευρώπη. Όσο ποτέ στο παρελθόν. Τι θα είδα λοιπόν συγκεκριμένα να κάνετε. σε ό,τι αφορά και την ε, πολιτική λιτότητα, η οποία μεταξύ άλλων και από εσά υποστηρίχθηκε. Πώς μπορεί να μειωθεί λοιπόν το χάσμα αυτό και πώς μπορεί να υπάρξει μια κοινωνική Ευρώπη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό για τον κόσμο για να υποστηρίξει την Ευρώπη. Και κατά δεύτερον, δεν θα σας προκαλέσει η έκπληξη του γεγονός ότι αν ε, σωστά καταλάβαμε σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις Ευρωπαίων Υπουργών Ιστορικών ε, θα υπάρξουν αυξημένοι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης ε, σε ό,τι αφορά την Frontex. Τι θέλετε να κάνετε λοιπόν για να διαμορφώσετε και να εφαρμόσετε μια ανθρώπινη πολιτική μετανάστευσης και πώς οι χιλιάδες που ξεβράζουν στις ακτές μας, ε, στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, θα μπορέσουν να βοηθηθούν με μια ανθρωπιστική πολιτική μετανάστευση. Νομίζω ότι ήταν αυτή μια από τις σημαντικότερες αξιώσεις των τελευταίων ετών. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Στο Μανώλη Γλέζο θα δώσουμε το λόγο που είναι και ο πρεσβύτερος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Σε αντιπροσωπεία ΣΥΡΙΖΑ που εξαπλασιάστηκε από τις προηγούμενες ευρωπαϊκές εκλογές. Ε, αγαπητέ Ζαν Κλοντ Γιούγκερ, θα ήθελα να ξέρω προσωπικά και η αντιπροσωπεία μας εάν γνωρίζετε ότι στην Ευρώπη όλοι ταυτίζεται η Κομισιόν το Διευθυντήριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τέτοιο σημείο ώστε να υπάρχουν και πολιτικοί οργανισμοί που να ζητούν να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέτοια είναι η ταύτιση που γίνεται. Και ρωτώ, εφόσον υπάρχει αυτό το θέμα της ταύτισης, η Κομισιόν θέλει την Ευρώπη των λαών ή την Ευρώπη του χρήματος. Θέλει την Ευρώπη της λαϊκής κυριαρχίας ή την Ευρώπη των μονοπωλίων και των ολιγοπωλίων. Θέλει την Ευρώπη των εκμεταλλευτών ή την Ευρώπη των εκμεταλλευομένων που ζητούν το δίκιο τους. Με μια γενική λέξη θα υπερασπιστεί το δίκαιο ή ναι ή όχι. Και όσον αφορά το κυπριακό θα ήθελα να πω είναι ανεπίτρεπτο εδάφη ευρωπαϊκά να βρίσκονται κάτω από την κατοχή τουρκικών στρατευμάτων εισβολής παρά τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τι θα κάνετε γι' αυτό. Και τελευταία, τελευταίο, η συμπεριφορά ως προς την Ελλάδα θα αλλάξει ναι ή όχι. Θα μας θεωρείτε ότι είμαστε μονάχα ένας χώρος θέρετρο, δηλαδή ένα ξενοδοχείο για όλη την Ευρώπη ή θα μας αφήσετε να αναπτύξουμε και την αγροτική μας οικονομία και την βαριά βιομηχανία και όλες τις, την αξιοποίηση των ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Vielen Dank, Manolis. Και τώρα το λόγο έχει ο Ντένις Ντεγιόγκ και μετά ο Ζωάο Φαρέρα. Uh, Ευχαριστώ Γκάμπη. Θέλω να καλωσορίσω τον Ζαν ε, Κλοντ και να του υποβάλω δύο ερωτήσεις για τα θέματα διαφάνειας. Το πρώτο αφορά το μητρό διαφάνειας ε, για τους ε, λομπίστες. Νομίζω ότι στους πρασίνους δηλώσατε ότι είστε υπέρ ενός υποχρεωτικού μητρώου. Αυτό νομίζω ότι είναι ευπρόσδεκτο για τη δική μας και για τη δική μας πολιτική ομάδα. Όμως, ερώτηση, θα υποβάλλετε πρόταση οι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι να μην λαμβάνουν, να μην δέχονται επισκέψεις από μη καταγεγραμμένους σε αυτό το μητρό λομπίστες. Δεύτερον, τελευταίο ερώτημα πάντα για τη διαφάνεια. Τα τελευταία χρόνια Είχαμε έναν πολύ επικοδομητικό διάλογο νομίζω με τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Σεύκοβιτς, για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων, expert groups, που η σύνθεσή τους ε, ήταν πάρα πολύ δυσανάλογη, κυρίως εκπροσωπούνταν ε, πολυεθνικές σε αυτά τα groups και ήθελε και ο αντιπρόεδρος Εύκοβιτς να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Βλέπουμε όμως ε, ότι και από τη Γενική Γραμματεία, Γραμματεία συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, επειδή είναι ανεξάρτητες οι γενικές διευθύνσεις να οργανωθεί κάτι τέτοιο. Ερώτηση λοιπόν, θα ενισχύσατε τη θέση του Γενικού Γραμματέα σε ό,τι αφορά τις γενικές διευθύνσεις, ώστε να μπορεί δηλαδή να υπάρχει ένας διάλογος ε, κυρίως με το Γενικό Γραμματέα. Και επίσης θα ήσασταν πρόθυμος ε, ενίοτε, φυσικά και ξέρω ότι δεν μπορείτε σε εβδομαδιαία βάση να το κάνετε, ίσως όμως κάποιες φορές το χρόνο θα ήσασταν ε, διατεθειμένος να έρχεστε σε επαφή με το intergroup που ελπίζω να συγκροτήσουμε για το θέμα αυτό εμείς και να μας ενημερώνετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ντένις Δε Γιόγκ. Ο Ζωάτορα. ευχαριστώ Γκάμπι. Γκάμπι, ευχαριστώ. Κύριε Γιόγκερ. Η κατάσταση στην Πορτογαλία, στη χώρα μου, δεν ε, είναι ε, μεμονωμένη αλλά είναι υποδειγματική, χαρακτηριστική. Μετά από ε, τις τρεις, ε, τρία χρόνια παρέμβαση στη Τρόικα που υποστηρίξατε βρίσκεται αντιμέτωπη η Πορτογαλία με τη μακρύτερη ύφεση που γνώρισε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Διαρθρωτική ανεργία που έχει εκτιναχθεί σε επίπεδα που δεν υπήρχαν ποτέ σε δημοκρατικά πολιτεύματα. Το ίδιο ισχύει για την ένδια τα τελευταία 40 χρόνια χρόνια. Ε, πρέπει να πέσουμε πίσω στα σκοτεινά χρόνια του φασισμού για να απαντήσουμε μια ε, αντίστοιχη κοινωνική κατάσταση. Κύριε Γιόνκερ, τι μπορούμε να πούμε ε, στους ανέργους, στους νέους, στους συνταξιούχους, στους εργαζομένους που περιμένουν περισσότερα από μας και από εσά από την ενιαία ψηφιακή αγορά ή το να μπορούν να μιλάνε στο κινητό χωρίς να πληρώνουν πληρώνουν την περιαγωγή. Θέλουν μισθό, θέλουν σύνταξη, θέλουν αξιοπρεπή ζωή. Θα ήθελα τώρα να ευθύσω την προσοχή σας σε δύο ζητήματα. Πρώτον, ε, έχει καταστραφεί, καταρακωθεί η οικονομία, είναι παροχημένα τα οικονομικά συστήματα, τα επενδυτικά επίπεδα έχουν πέσει στα επίπεδα της δεκαετίας του 50, του προηγούμενου αιώνα και τώρα για το χρέος ε, ε, έχει ξεπεράσει το 30% του ΑΕΠ και το ή... 21 εκατομμύρια ε, θα φεύγουν από τη χώρα ε, και ε, την ημέρα αν δεν αλλάξουμε την κατάσταση. Και θα ήθελα ε, να σας ρωτήσω το εξής. Ε, προτίθεστε να δεχθείτε την αναγκαιότητα της επαναδιαπραγμάτευσης ε, του δημοσίου χρέους σε χώρες όπως η Πορτογαλία. Μιλάω για τα επιτόκια, για τις προθεσμίες αποπληρωμής, για το επίπεδο του χρέους, ούτως ώστε να συμβαδίσει επιτέλους με τις αναπτυξιακές ανάγκες το χρέος. Και δεύτερον, και κλείνω, Αναγνωρίζει, ε, αναγνωρίζεται κύριε Γιούγκερ την ανάγκη να προσαρμοστεί το καθεστώς του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα κάνω μια διακοπή γιατί θέλω να κλείσετε το κινητό σας και να με ακούσετε. Η γυναίκα μου ήταν, απαντάει ο κύριος Γιούγκερ. Η δεύτερη ερώτηση που θέλω να σας κάνω ξέρω να κάνω και δύο πράγματα ταυτόχρονα. Μπορώ να σας ακούω και να γράφω ε, ότι όλα πάνε καλά. Καταλαβαίνετε και πορτογαλικά, γιατί εγώ περιμένω να βάλει τα ακουστικά για να καταλαβαίνετε και τι λέω. Ε, μεγάλωσα στα νότια προάστια του Λουξεμβούργου. Σχεδόν όλοι οι γειτονές μου Πορτογάλοι ήταν. Ε, ξέρω πάρα πολλά για την ε, ε, Πορτογαλία, μην ανησυχείτε. Πολύ ωραία, συνεχίζει ο κ. Φερέιρα. Η δεύτερη ερώτησή μου είναι η εξής. Ε, ε, αναγνωρίζετε ε, μέσα σε αυτό το πρόγραμμα που είχατε ευγενή καλοσύνη να μα στείλετε την αναγκαιότητα προσαρμογής του καθεστώτος του Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με τον πληθυσμό του. Εννοώ το καθεστώ και τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και ρωτάω εάν μια χώρα της Ευρωζώνης τελικά αποδειχθεί ότι δεν μπορεί με βιώσιμο τρόπο να παραμείνει στην Ευρωζώνη και πρέπει να ανακτήσει την κυριαρχία της σε νομισματικό και δημοσιονομικό επίπεδο. Είστε διατεθειμένος να δεχθείτε ε, το ενδεχόμενο μιας διαπραγματευμένης εξόδου από την Ευρωζώνη μιας χώρας ε, που θα έχει την επιτακτική ανάγκη να το κάνει για να υπερασπιστεί το μέλλον της και την οικονομία της. Σας ευχαριστώ και σένα, Ζωάη. Αγαπητοί φίλοι, σας παρακαλώ, μία-δύο ερωτήσεις αναομιλητή. ιδάλος. Ήταν μεγάλη εισαγωγή. Θέλουμε να λάβουμε και μία απάντηση από τον κύριο Γιούγκερ. Τώρα λοιπόν ε, σας πετάω το μπαλάκι κύριε Γιούγκερ και να σας ζητήσω να περιοριστείτε σε πέντε λεπτά. Πολύ λυπάμαι. Αλλά η δεν θα καταφέρουμε. 15 ερωτήσεις ε, μου θέσατε και μου ζητείτε να δώσω μια απάντηση μέσα σε 5 λεπτά. Αυτό χαρακτηρίζει την ποιότητα του δημοκρατικού διοργανικού διαλόγου. Ξέρετε, δεν είμαστε στην τηλεόραση. Ε, στην τηλεόραση είχαμε μετριότατες, θα έλεγα, θλιβερές συζητήσεις. Ε, καλό θα ήταν εδώ να είναι κάπως διαφορετικό ε, το πράγμα, να μπορούμε να αφιερώσουμε τη δέουσα σημασία στα πολύ σημαντικά αυτά ευρωπαϊκά θέματα. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να απαντήσω στο πόδι ε, βιαστικά γιατί κάθε ε, θέμα ε, απαιτεί μια απάντηση. Περνάω στα γερμανικά τώρα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι και εδώ πέρα συνεχίζονται τα πράγματα όπως πριν. Απλά συνεχίζεται η κατάσταση. Αλλά αυτό δεν είναι. Δεν μπορεί ούτε εδώ ούτε αλλού να συνεχίσουν τα πράγματα όπως ήταν. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουν τα πράγματα και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι όπως ε, τα πηγαίναμε. Ναι. Και συνεχίζω στα γαλλικά. Ε, πρέπει να έχετε υπόψη σας ε, σε ποιον μιλάτε για να μην πω πρέπει να σας ρωτήσω ποιοι, είστε, νομίζετε ότι είστε και σε ποιον νομίζετε ότι απευθύνεστε. Τι είμαι εγώ, είμαι γιος κανενός εκατομμυριούχου που ε, γεννήθηκα σε χρυσή κουνιά. Εκεί με κοίμιζαν οι γονεί μου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα και ποτέ δεν θα δεχθώ να έχουμε τους καλούς και τους αγίους, τους αποστόλους από τη μία πλευρά ε, που κάνουν θαύματα μόνο και από την άλλη να έχουμε τους βρωμερούς καπιταλιστές σαν και εμένα. Δεν μπορώ να το δεχθώ. Και από την άλλη πλευρά, κύριε, εγώ δεν πιέζομαι να σας σεβαστώ, σας σέβομαι. Και σας παρακαλώ να πράξετε το ίδιο αν μπορείτε. Λοιπόν, ανέφερα και εγώ κάποια από τα προβλήματα τα οποία εσείς θίξατε είπανε ότι στην Ευρώπη ε, λίγο πολύ παντού υπάρχει αυτή η σύγχυση που γίνεται ε, μεταξύ Κομισιόν και Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ταυτίζεται με την Κομισιόν και το αντίστροφο. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι το ίδιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μικρότερη από την Ευρώπη. Τέλο πάντων, από εκεί και πέρα. Οι εφημερίδε, όλε οι εφημερίδε, όταν λαμβάνει μια απόφαση, προτείνει κάτι, παίρνει μια πρωτοβουλία η Κομισιόν, γράφουν εφημερίδε η Ευρώπη. Μα η Κομισιόν δεν είναι η Ευρώπη. Η Κομισιόν πρέπει να υπηρετεί το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών και η Κομισιόν από μόνη δεν μπορεί να ε, κάνει τίποτα να κινήσει Υπάρχουν ε, πάρα πολλοί άλλοι ε, που επηρεάζουν, πολιτικο-συνδικαλιστικοί φορείς και πολλοί άλλοι. Δεν μπορεί η Κομισιόν δηλαδή να τα κάνει όλα μόνη. Δεν μπορεί να γίνεται λοιπόν αυτή η ταύτιση μεταξύ Ευρώπης και Κομισιόν. Εμένα με ενδιαφέρει και το κοιτάζω καθημερινά και πάρα πολύ κοντά το τι γίνεται στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία, γιατί έχω και στις δύο χώρες πολλούς φίλους. Και όταν διατελούσα, όταν ετέλεσα πρόεδρος ε, του Eurogroup της Ευρωομάδας, ε, τότε τηλεφωνούσα τρεις φορές τη μέρα σε μάρτυρες, σε αυτό, μάρτυρες από το δρόμο, στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, για να... Δεν θέλω να το πω με απλουστευτικό τρόπο. Για να πάρω το σφιγμό τέλος πάντων ε, και ξέρω ε, τι εκτροπές ε, και τι διολυστήσεις υπήρξαν. Αλλά θα πρέπει να λάβετε υπόψη πρώτον ότι η κατάσταση στις χώρες αυτές δεν... Πώς να το πω... Δεν δημιουργήθηκε δεν κόπηκε και ράφτηκε από την Ευρώπη και επίσης ότι εμείς βλέπαμε τι γίνεται. Π.χ. έρχομαι στη διαφθορά. Υπάρχει ε, παράδοση σε κάποιες χώρες. Δεν θα ούτε ήμουν εγώ αυτός που θα απαγόρευε ή απαγόρευσε στους Έλληνες, ελληνικές αρχές να φορολογούν τους πλούσιους, τους ονάσιδες και τους άλλους. Ούτε ήμουν εγώ αυτό που υποχρέωσε ή που έφερε τι αρχέ στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία να μειώσουν τον κατώτατο μισθό και μάλιστα το αντίθετο ε, υποστήριζα. Κάποιε χώρε που ε, είναι φτωχέ με εξέπληξε το ότι ε, απαιτούσαν να γίνουν αυτές οι πολιτικές, ζητούσαν από τα εθνικά κοινοβούλια βοήθεια. Χώρες όπως η Πορτογαλία, όπως η Ελλάδα φτωχές που είχαν χαμηλά, πολύ μικρά προνοιακά επιδόματα. Είναι πολύ δύσκολο και πολύ πλοκό το τοπίο. Δεν μπορούμε να τα βλέπουμε όλα έτσι χωρίς να γνωρίζουμε τόσο καλά την κατάσταση και την κοινωνική κατάσταση σε ορισμένες χώρες. Εγώ πιστεύω ότι στην Ευρώπη πρέπει σε αυτό το τοπίο το κατακαιρματισμένο να δώσουμε μια απάντηση. Και έρχομαι στο θέμα της μετανάστευσης και της νόμιμης μετανάστευσης. Ε, εξευρωπαϊσμός, αν θέλετε, η ευρωπαϊκοποίηση χωρίς εναρμόνιση όμως του δικαιώματος ασύλου. Η παράνομη λαθρομετανάστευση είναι ένα πρόβλημα και ναι είμαι υπέρ της ενίσχυσης τη προστασία των εξωτερικών συνόρων, διότι αυτοί οι οποίοι πήγαν να ψηφίσουν στις 25 Μαΐου και ψήφισαν κατά της Ευρώπης, πολλοί εξ αυτών το έκαναν μεταξύ άλλων γιατί νομίζουν ότι δεν του προστατεύει επαρκώς η Ευρώπη ή τους προστατεύει ανεπαρκώς. Επομένως, ε, ο Frontex ε, που έχει ένα προπολογισμό γελίο των 80 εκατομμυρίων ε, πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο για να μπορεί να καταπολεμήσει την ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση. Θα ήθελα όμως να σας απευθύνω μια έκκληση. Είναι σκανδαλώδες οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες να μειώνουν ε, τις ε, δημόσιες ε, αναπτυξιακές ενισχύσεις, να αναθεωρούν επιταχύρω προς τα κάτω τα ποσά, να μην... επενδύουν παρά εκεί που πραγματικά χρειάζεται. Υπάρχουν τρεις ή τέσσερις χώρες που αντιστοιχούν στα κριτήρια της αναπτυξιακής βοήθειας. Υπάρχει μια αδικία, βαρύτατη αδικία, η οποία γίνεται και που έχει ως αποτέλεσμα αυτοί που δεν μπορούν να ζήσουν στις χώρες τους, παίρνουν ε, ένα σκάφος ή μην μπαίνουν σε μια σχεδία για να φτάσουν στην Ιταλία ή στην Ελλάδα να βρουν μια καλύτερη μοίρα. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες να ε, σταθούν στα πόδια τους, ε, να στήσουν την οικονομία στα πόδια τους και να αλλάξει ε, όρους του χρήματος. Δηλαδή όχι να αγνοούμε ε, τις χώρες από τις οποίες εκεί ξεκινάει εξαθλίως και να μην δίνουμε αναπτυξιακή βοηθεία. Εγώ λοιπόν είμαι υπέρ μιας ε, αύξησης της αναπτυξιακής βοήθειας, να δίνεται με μεγαλύτερη συνέπεια και λογική και επίσης στην Ιταλία, στην Ελλάδα, όπου χρειάζεται. Καλό θα ήταν να υπάρξουν γραφεία για τους πρόσφυγες και οι βόρειες χώρες θα έπρεπε να είναι πιο αλληλέγγυες απέναντι στις νότιες. Λέμε Mare Nostrum τη Μεσόγειο. Δεν είναι όμως ε, η θάλασσα του Νότου. Πρέπει να υπάρξει ε, πραγματικά μεγαλύτερη συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ Βορρά και Νότου ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των συνεπειών της ανεξέλεγκτης λαθρομετανάστευσης. Το πρόβλημα του ασύλου. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε από κοντά ώστε όσο είναι δυνατόν να εξαλείψουμε αυτές τις ε, μεγάλες διαφορές από τη μια νομοθεσία στην άλλη. Ο ίδιος φάκελος που υποβάλλει το ίδιο άτομο σε μία χώρα μπορεί να έχει 80 ή 90% δυνατότητες να εγκριθεί και σε μια άλλη 1% ε, πιθανότητες να εγκριθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικά λοιπόν όλα αυτά. Και θα πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτά. Τώρα, σε ερωτήσεις που αφορούν την Ισπανία συγκεκριμένα δεν μπορώ να απαντήσω. Γνωρίζω ότι η Ισπανία είναι μια μεγάλη χώρα, η Ευρώπη όμως είναι, ε, δεν είναι Ισπανία. Ε, είναι το δικαίωμα της απεργίας ε, μεταξύ όλων των άλλων εθνικό και ευτυχώς οι εθνικοί νομοθέτες καταφέρνουν σε ό,τι αφορά κάποιες διατάξεις της νομοθεσίας να τις διατηρούν ευνοϊκές προς για την μη τήρηση, για το μη σεβασμό του δικαιώματος της απεργίας ή για το πρόβλημα με την άμβλωση είναι θέματα πολύ σοβαρά. Δεν μπορούμε να τα εξετάσουμε εδώ ακροθυγώς. Πιστεύω ότι θα πρέπει οι εθνικές αρχές, αυτές που είναι αρμόδιες να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα τα εθνικά, με την απεργία, με την άμπλης. Τώρα, για τη διαφάνεια. Είμαι της άποψης ότι το μητρό, η τα μητρώα ε, ανθρώπων που συμμετέχουν σε ομάδες λόμπι ε, πρέπει να είναι δημόσια. Να ξέρουμε ποιος ε, ανήκει στην κατηγορία του λομπίστα ή όχι. Τώρα το να μην ε, να ζητήσουμε από τα στελέχη της δίκησης να μην δέχονται στο γραφείο τους ε, ένα λομπίστα ή όχι, είναι δύσκολο. Μπορεί εσείς να μην είστε σε μια λίστα ε, λομπίστα, ε, πώς θα μπορεί να απαγορεύσει κάποιος σε ένα στέλεχος της δίκησης να δεχθεί κάποιους ανθρώπους στο γραφείο του. Η Επίτροπη και ο πρόεδρος συναντώνται με πολλούς. Απλά πρέπει να λένε με ποιους συναντώνται. Από τις τράπεζες, από τις ε, πολυεθνικές, από οπουδήποτε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια διοργανική ρύθμιση, ένας διοργανικός διακανονισμός σε όλα τα θεσμικά όργανα για να έχουμε τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια για αυτές τις ομάδες εμπειρογνωμόνων ε, που ε, αναπτύσσονται και πληθαίνουν ε, στους κύκλους της Κομισιόν. Να δούμε πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης μπορεί να συμμετέχει περισσότερο στη στελέχωση αυτών των ομάδων. Ίσως οι βουλευτές θα έπρεπε να έρχονται αυτοπροσώπως στις συνεδριάσεις αυτών των ομάδων εμπειρογνωμών, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, ναι μεν προσκαλούνται, αλλά δεν έρχονταν και έστελαν κάποιον άλλον στη θέση τους. σε ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα να διαβάσω τον ε, κατάλογο των επόμενων πέντε ομιλητών. Για να είσαστε προετοιμασμένοι και να μην ανησυχείτε. Γιώργ. Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli und Pablo Iglesias. Uh, ναι, είμαι η Μάλιν Μπιόρκ από το αριστερό κόμμα της Σουηδίας ε, και θα ήθελα μόνο να πω ότι συμφωνώ με τους συναδέλφους ε, που έθεσαν τα ζητήματα της πολιτικής της Τρόικα και πώς αυτό συνέβαλε στην διόγκωση των ανισοτήτων ε, στις χώρες αλλά και ανάμεσα σε χώρες είναι μια ανάλυση, ένα γεγονός, ένα δεδομένο ε, το οποίο ε, ε, δεχόμαστε κι εμείς και προέρχομαι από βόρεια χώρα. Θα ήθελα τώρα, στα πλαίσια των ερωτήσεων, αν εκλεγείτε πρόεδρος, να επικεντρωθώ στο θέμα της ισότητας των δύο φύλων. Νομίζω ότι εκεί παρουσιάζονται μεγαλύτερες ελλείψεις. Η φτώχεια είναι γένους θηλυκού σήμερα και βλέπουμε τα προβλήματα των μεταναστριών. Μία στις τρεις γυναίκες πάνω από τα 15 έχει υποστεί ε, σωματική ή ψυχολογική βία. Οπότε θα ήθελα να σας θέσω μια άμεση ερώτηση με ποιο τρόπο θα εξασφαλίσετε μεγαλύτερη ισότητα των δύο φύλων αν εκλεγείτε η, επόμενη χρονιά που είναι τα 20 χρόνια από την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου ε, υπολείπονται όλοι οι στόχοι με ποια δράση θα αναλάβετε και θα αναλάβετε επίσης νομική δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Σας ευχαριστούμε Μάλιν. Ε, ήσασταν και σύντομοι όπως σας ζήτησα. Η Μαρτίν Άντερσον τώρα. Μάρτιν Άντερσον από το Sinn στην Ιρλανδία. Υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα που θέλουμε να θέσουμε σε σχέση με την Ιρλανδία. Πρώτον, τι θα γίνει με την Ιρλανδική ειρηνευτική ε, διαδικασία και δεύτερον, το οικονομικό ζήτημα και ο, θα το ε, σχολιάσει αυτό. Όταν η εκτελεστική κυβέρνηση συγκροτήθηκε στην Βόρεια Ιρλανδία, ο πρόεδρος Μπαρόζο ε, συνέβαλε συστήνοντας ε, μία task force για να επικουρήσει την κοινή κυβέρνηση ΣΥΝΦΕΝ και UDP ε, στο δρόμο τους προς την Ευρώπη. Προέκυψαν δυσκολίες και αυτή τη στιγμή υπάρχουν εσωτερικές δυσκολίες που δεν θα σχολιάσω, δεν θα αναφέρω εδώ σήμερα. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω εάν θα συνεχίσετε με αυτή την Task Force για τη Βόρεια Ιρλανδία και δεύτερον ο Μάρτιν Μαγκίνες, ο, ο κοινός πρωθυπουργός, ε, θα έρθει ε, στις 22 του μήνα. Ε, εάν έρθει θα τον συναντήσετε, ούτω ώστε να ενημερωθείτε εκ των έσω για τα όσα συμβαίνουν στα πλαίσια της ενευτικής διαδικασίας. Ευχαριστώ, Μιρόσλαφ Ράνστολ. Bonjour, Monsieur Juncker. <coughs> Κύριε Juncker. Λυπούμε γιατί δεν μιλήσατε λουξεμβουργιανά. Δεν μιλήσατε τη διασκεδαστική αυτή γλώσσα. Ε, Εμένα μου αρέσουν τα λουξεμβουργιανά, λέει στα λουξεμβουργιανά και ο συνάδελφος. Εγώ θυμάμαι ότι Όταν ε, ήσασταν πρόεδρος του Eurogroup, ε, δουλέψατε με μεγάλη αξιοπρέπεια και στηρίξατε και την επέτειο ε, της ανόδου της δυναστείας του Λουξεμβούργου στον τσεχικό θρόνο το 2010. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμβουλή αυτή. Τέλος πάντων, να έρθω τώρα σε ένα ερώτημα. που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Σε ποιο βαθμό ή μάλλον τι μέτρα θα μπορούσατε να λάβετε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σταθεροποίηση της Ευρωζώνης. Διότι υπάρχει μια πολύ σοβαρή κατάσταση με την νομισματική κρίση που υπάρχει και θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί κατεπηγόντως το πρόβλημα. Äh, Σας ευχαριστώ Μυροσλάφ. Και τώρα η Μπαρμπάρα Σπινέλη έχει το λόγο. Θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα στον κύριο Γιούγκερ. Ποια θα είναι πραγματικά τα σημεία τα οποία θα αλλάξετε σε σχέση με την προηγούμενη ε, επιτροπή και σε ό,τι αφορά την Τρόικα. Είπατε ότι το εργαλείο αυτό θα το εγκαταλείψετε, θα το αφήσετε. Η Τρόικα με τι θα αντικατασταθεί λοιπόν στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά τώρα το δεύτερο σημείο, την ευελιξία την ευελιξία και την ε, απαραίτητη βελτίωση του μέσου αυτού. Μία αλλαγή στην πολιτική θα μπορούσε να περιλαμβάνει αλλαγή των επενδυτικών ε, σχεδίων σε ό,τι αφορά και τα σχετικά ε, μέσα. Ένα οικονομικό New Deal με κοινωτικά μέσα. Ύστερα, σε ό,τι αφορά τον ε, Επίτροπο για τη Μετανάστευση, θα υπάρχει τέτοιος Επίτροπος με πραγματικές, ουσιαστικές εξουσίες. Με εξουσίες που θα συνενώνουν ευθύνες και δικαιοσύνης αλλά και εσωτερικών υποθέσεων. Ναι, ναι, να μην υπάρχει δηλαδή μόνο ένας ε, επίτροπος όπως η Μάλμστρομ η οποία έλεγε «Ε, έχουμε, δεν έχουμε λεφτά για να σώσουμε τον κόσμο που πεθαίνει στη Μεσόγειο. Ευχαριστώ πολύ». Ευχαριστώ όλοι, Πάρμαρα λέει η πρόεδρος, ο Πάμπλο Ιγκλέζης έχει τώρα το λόγο. Από το Ποδέμος, Παύλο ε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γιούγκερ που είστε εδώ. Πιστεύω ότι η παρουσία σας, ε, η διάθεσή σας να συζητήσετε μαζί μας λαμβάνοντας υπόψη ε, ότι ήδη έχετε εξασφαλίσει τη στήριξη των ε, συντηρητικών και των σοσιαλιστών, το ότι έρχεστε εδώ είναι σημαντικό, είναι αξιέπαινο. Πρέπει να σας πω όμως ότι εμείς εδώ κύριε Γιούνκερ δεν ε, μπορούμε να συνεχίσουμε να επιβραβεύουμε τους ε, κλέφτες και τους απατεώνες. Και πραγματικά κρούμε τον κόδωνα ε, του κινδύνου ε, στις χώρες του Νότου. Αν εσείς είστε ε, στα ενία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήσασταν πρωθυπουργός ενός φορολογικού παραδείσου του Λουξεμβούργου. Μιλάτε για κατώτατο μισθό. Καλό αυτό, αλλά οι πολιτικές λιτότητας που εφάρμοσε και εφαρμόζει η Τρόικα και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, τι αποτέλεσμα έχουν ο κατώτατος επαγγελματικός μισθός στη χώρα μου να είναι 645 ευρώ το μήνα και η κατάσταση στην Πορτογαλία ή στην Ελλάδα να είναι ακόμα χειρότερη. Πολύ καλό είναι που λέτε ότι δεν, έρχεστε, ε, δεν κατάγεστε από οικογένεια εκατομμυριούχων ε, ή ότι είχατε κι εσείς υπάρξει συνδικαλιστής, αλλά σε μια γερμανική εφημερίδα Λέω ότι δώσατε μία ε, συνένταξη ε, για μία, σε μία συνομοσπονδική γερμανική εταιρεία ασφάλειας κτλ. Και, και πήρατε 15.000 ευρώ για αυτή την παρουσίαση έχουν εξαφανιστεί 5,8 εκατομμύρια ευρώ από, ε, σε φορολογικούς παραδείσους που θα μπορούσαν να πάνε σε σχολεία και σε ε, νοσοκομεία. Εμένα μου αρέσει ε, και κάποιο να είναι αυστηρός και να λαμβάνει αποφάσεις. Να είναι αυστηρός όμως ε, ενάντια στους ισχυρού και όχι στους αδύναμους, στους ανίσχυρους. Ρωτώ λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα κάνετε, θα προωθήσετε τη μεταρρύθμιση των ε, ποινικών θεσμών στις χώρες της ώστε οι φοροφυγάδε να μπαίνουν στη φυλακή ακόμη και αν αυτό μπορεί να αφορά κάποιες ε, έτσι, εξέχουσες προσωπικότητες της Ένωσης. Σας ευχαριστώ και έτσι θα κλείσουμε τον ε, γύρο αυτό. Σας δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Καλά τα λέτε κύριε Ιγκλέσιας. Θυμήσατε ότι η χώρα από την οποία προέρχομαι έχει τον υψηλότερο ε, κατώτερο μισθό ε, στην Ευρώπη, ε, το υψηλότερο ελάχιστο εισόδημα στην Ευρώπη, τις υψηλότερες οικογενειακές παροχές και έχετε δίκιο όταν υπενθυμίζετε τη σχέση με τα εισοδήματα στον τρίτο κόσμο. Ναι, ε, είναι αληθή αυτά που λέτε, όμως είναι πολύ σύντομη η παρέμβαση και δεν μπορώ να επεκταθώ. Ε, όταν είχαμε λάβει την Προεδρία, εγκρίθηκε κώδικας και διοντολογίες από το ε, Συμβούλιο σε σχέση με ε, με τα φορολογικά ζητήματα. Εγώ ίδιος ε, κατήργησα το τραπεζικό απόρριτο και με, ε, υπάρχει η πρόθεση να αλλάξει η κατάσταση και με, είπατε ότι στον τομέα των επιχειρήσεων ε, θα πρέπει να υλοποιήσουμε αυτό που είπαμε για την εκείνη φορολογική βάση και δεν μπορούσατε να κρύψετε και τη χαρά σας. Ε, κοιτάξτε, θα πρέπει εκεί πέρα που παράγεται το κέρδος, εκεί και να φορολογείτε. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Ε, σε κάθε περίπτωση έχετε στη διάθεσή σας ε, πάρα πολύ εκτενείς πληροφορίες σε σχέση με άλλους. Ε, το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο σε αυτό το τομέα δεν υπάρχει ή τουλάχιστον όχι ε, σε μεγάλη κλίμακα και η καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής ε, αλλά και τα ζητήματα ποινικού δικαίου ε, θα πρέπει ε, σταδιακά μόνο να αντιμετωπιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε σχέση τώρα με την ασφάλεια θα ήθελα να σας πω ότι Σε επίπεδο ε, πληθυσμού, το πρόβλημα της διατροφικής ασφάλειας, ε, το πρόβλημα της ε, φτώχειας δεν απαιτεί μία στρατιωτικού χαρακτήρα απάντηση. Χρειάζεται soft power να αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο την διπλωματική οδό και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τα συμπεράσματα του ε, Συμβουλίου σχετικά ε, του Δεκεμβρίου σχετικά με αυτό το ζήτημα. Δεν ξέρουμε τι πρέπει να αντικαταστήσουμε την Τρόικα. Δεν έχω έτοιμη την απάντηση. Χρειαζόμαστε ε, ένα πιο ενάρετο εργαλείο, ένα δημοκρατικότερο εργαλείο στη θέση της Νομίζετε ότι θέλει να είναι τόσο ε, εμπνευσμένο ένα δημοκράτη που να μιλάει για τέτοιε αρετέ. Δεν ισχύει αυτό. Μίλαγα για τη δημοκρατική αρετή. Είναι αρετή η δημοκρατία. Αυτό εννοούσα. Η Τρόικα ε, πρέπει να νομιμοποιηθεί από σε πλευρά προς το παρόν δεν νομιμοποιείται δημοκρατικά. Θα δούμε με ποιο όργανο θα την αντικαταστήσουμε. Αν θεωρείτε ότι ο καλύτερος τρόπος για να καταπολεμήσουμε τα ελλείμματα είναι να δημιουργήσουμε νέα ή για να καταπολεμήσουμε το χρέος πρέπει να το αυξήσουμε, δεν ε, μπορούμε να καταλήξουμε σε κάτι που θα περιγράφαμε ε, κοινέ ε, απόψεις. Εγώ είμαι αλλεργικός στο δημόσιο χρέος και θεωρώ ότι ε, απατώνται όλοι όσοι ε, προκρίνουν αυτή την οδό διότι θα πληρώσουν τα σπασμένα η φτωχή του μέλλοντος. Ε, χρειαζόμαστε σταθεροποίηση της Ευρωζώνης. Ναι, ναι, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και στην Τραπεζική Ένωση, διότι σπάμε τα δεσμά ανάμεσα στις τράπεζες και στα δημόσια χρέη. Ε, σταθεροποίηση λοιπόν της Ευρωζώνης. Τι σημαίνει αυτό ότι θα καταραστούμε όλους όσους έχουν δημοσιονομικά προβλήματα και δημιουργούν δυσκολίες ε, στους υπόλοιπους. Όχι, πρέπει να ε, βοηθήσουμε και να σεβαστούμε τις χώρες προγράμματος, όχι να τις καταραζόμαστε. Και δεν θέλω τώρα για το ευρώ και για τα προγράμματα των διαφόρων χωρών να ανοίξουμε αυτή τη στιγμή συζήτηση, αλλά ε, η κάθε συζήτηση θα πρέπει να προσαρμοστεί στην ιδιαίτερη κατάσταση που επικρατεί σε κάθε χώρα. Οπότε, όταν μιλάμε για την Ευρωζώνη, θα πρέπει ταυτόχρονα να λαμβάνουμε υπόψη τις κυβερνήσεις αλλά και τους λαούς ε, της Ευρώπης ε, και να υπάρξει σεβασμός όλων προς όλους για όλα τα συναφή ζητήματα αυτού ε, του διπόλου, δηλαδή μιλάω για την ισότητα των δύο φύλων, ε, απευθύνθηκα ήδη στις κυβερνήσεις, ούτως ώστε να υπάρχει ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα, Εγώ ως επίτροπο πρότεινα για 15 χρόνια γυναίκα και Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει μία λιγότερη γυναίκα σύνθεση της Επιτροπής αυτή τη φορά, αλλά σίγουρα πρέπει να γίνει σεβαστή ε, όχι μόνο η ποσόστοση, η σημασία που έχουν οι γυναίκες ε, στην πολιτική ζωή. Δεν θέλουμε ένα... Μια λέσχη αντρών. Δεν θέλουμε να γίνει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, αλλά αυτό είναι απόφαση των κυβερνήσεων για την ισότητα των δύο φύλων πέρα από την πτυχή ε, διακριτικής μεταχείρισης δεν βλέπω πώς θα μπορούσε να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πάλι εδώ διότι ε, είμαστε δεσμευμένοι από το οικογενειακό δίκαιο και εν μέρει και από το αστικό δίκαιο των κρατών μελών. Δεν Απορρίπτουμε την διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ε, ε, λόγω φύλου, αλλά δεν ε, βλέπω με ποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να νομοθετήσει σε αυτό τον τομέα κάθε φορά που μιλάει για τη διακριτική μεταχείριση και προσπαθεί να κάνει τη φωνή της να ακούσει, ε, κυρίως στον τομέα της ε, οικογενειακής βίας που είναι μάστιγα στην Ευρώπη, προσκρούμε στο ίδιο κόλλημα ότι δεν είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα και οι εθνικοί νομοθέτες ε, πρέπει να αναλάβουν εκείνη οι διατάξεις. Φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί με πυγμή να καταγγείλει τα προβλήματα και να τροφοδοτεί τη συζήτηση σε εθνικό επίπεδο, αλλά μέχρι εκεί. Θα σταματήσω στο σημείο αυτό γιατί δεν μπορώ να συνεχίσω. Ναι, θέλω μόνο να μου κάνετε σήμα όταν έχετε ολοκληρώσει τις απαντήσεις σας. Όταν, όταν έτσι ε, κατηφορίζει, γιατί κλείνει η φωνή μου, τότε μπορείτε να συμπεραίνετε ότι κάθε φορά ότι ε, σταματάω. Μάλιστα, πολύ ωραία. Με τη φωνή δηλαδή να τα πάρουμε. Πολύ ωραία. Ο κύριος Μελανσόν. Γκάμπι, Γκάμπι, συγγνώμη, θέλω μία απάντηση σε ό,τι αφορά την Ιρλανδική διαδικασία. Ναι, δίκιο έχετε. Δίκιο έχετε η Ματίνα Άντερσον μου υποδεικνύει ότι έγινε συγκεκριμένη ερώτηση για την Ιρλανδική ειρηνευτική διαδικασία και σε ό,τι αφορά τη συνέχιση της Tax Force. Δύο ερωτήσεις. Ε, συγγνώμη, ξέχασα την πρώτη και της έλεγα να μου υπενθυμίσει την πρώτη. Η δεύτερη, σε ό,τι αφορά την Ιρλανδία, εγώ σκοπεύω να συνεχίσω αυτά που γίνονται. Και δεν έχω χρόνο στις 21 Ιουλίου να συναντηθώ με τον συνάδελφο που αναφέρατε. Δεν θα είμαι στις Βρεξέλλες την ημερομηνία αυτή. Είναι εθνική αργία αυτό, ξέρετε, στο Βέλγιο. Ερώτηση εκτός μικροφώνου, σχόλιο. Μάλιστα. Ωραία, λέει η πρόεδρος. Θέλετε να συνεχίσετε, μάλιστα. Πολύ ωραία. Ζωάν Λεκ Μελανσόν και μετά ο Νεοκλής. Μερία Κόιλεν, Άννα Χάζελχαμπ. Ε, Κύριε Γιούνκερ, καταρχάς ε, ε, να σας καθησυχάσω ότι αυτά που σας έχω φυλαγμένα που λέτε ότι δεν, σας, δεν καλά για σας δεν είναι συγκεκριμένα για σας όλα αυτά. Τέλος πάντων, το ότι ήρθατε εδώ είναι αξιέπαινο. Ε, δυστυχώς όμως το όνομά σας και η θέση σας ε, θα είναι συνώνυμο αυτά, αυτών που απεχθανόμαστε. Δηλαδή όταν είστε στην υπηρεσία των τραπεζών ε, και των καπιταλιστών δεν έρχομαι σε την παράθεση μαζί σας προσωπικά, έχετε την πλειοψηφία, ε, απεφάσισε ο Ευρωπαϊκός Λαός, ήρθατε εδώ να σας ε, ακούσουμε και να δούμε και το σε αυτή την τεράστια πόσα που μας χωρίζει. Εμείς δεν πιστεύαμε βέβαια ότι η κοινωνική προέλευση καθορίζει κάτι. Τώρα εμείς σας μιλάμε για την άμβλωση, μιλάτε για το οικογενειακό δίκαιο. Δεν νομίζουμε ότι αυτό έχει να κάνει. Ε, μιλάμε για τη μετανάστευση, μας απαντάτε για τη Frontex. Ενώ θέλουμε να σας πούμε ότι Υπάρχουν συμφωνίες με τις ε, χώρες ε, οι οποίες καταστρέφουν τις τοπικές τους οικονομίες. Τέλος πάντων, είστε ευφύς, θα είμαι πολύ συγκεκριμένος ε, στις δικές μου ερωτήσεις. Πρώτον, μεγάλη διατλαντική αγορά. Εσείς αναλαμβάνετε δεσμεύσεις, ας πούμε ότι σας πιστεύουμε. Δεν είναι όμως πρακτική της δημοκρατίας να πιστεύει μόνο αυτόν που αποφασίζει. Με ποιο τρόπο ο κόσμος, ο λαός θα μπορέσει να συμμετέχει στις διαβουλεύσεις όταν ε, φτάσει στην κατάσταση αυτή η συμφωνία προ υπογραφή, προ έγκριση. Ποιο θα το κάνει αυτό τα κοινοβούλια ή κάτι πολύ πιο τολμηρό θα μπορούσαμε να φανταστούμε ενδεχομένω λαϊκά δημοψηφίσματα. Ο κύριος ε, ε, Σνόουντεν ε, που άλλοτε φαίνεται ευεργέτης και άλλοτε ο τρομερός εχθρός. Είδαμε τι κάνει όμως η κατι πολυ πιο τολμηρο θα μπορουσαμε να φανταστουμε δεχομενως λαικα δημοψηφισματα ο κυριος σνοουντεν που αλλοτε φαινεται ευεργετης και πώς κατασκοπεύει. Τι θα κάνετε εσείς να μπορούν όχι μόνο ο κύριος Σνόουντεν αλλά και ο Αμερικανός πληροφοριοδότης να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Άλλα θέματα τα οποία αναφέραν και κάποιοι προλαλήσαντες. Δεν θέλω ε, να ε, στοχεύσω σε εσά και στη χώρα από την οποία κατάγεστε συγκεκριμένα. Σέβεστε τη χώρα μου, σέβομαι τη δική σα Παρόλα αυτά, το 2013 ακολουθεί η χώρα σα να συγκαταλέγετε στη λίστα με τους φορολογικούς παραδείσους. είναι, ποια είναι η πρώτη μάστιγα. Οι κλέφτε πηγαίνουν ε, στους φορολογικούς παραδείσους και κρύβουν εκεί τα λεφτά που τους έδεσαν οι πολίτες και τις τα πηγαίνουν τα χρήματά τους σε χώρες που ήδη είναι οι πιο πλούσιες. Μην το πάρετε προσωπικά, αλλά είναι λογικό ε, να σας κάνουμε αυτή την ερώτηση, γιατί ανήκετε σε μια χώρα που συμμετέχει σε αυτή τη βιομηχανία της κλοπής. Και επειδή μιλήσατε για την Ευρωπαϊκή Επικράτεια, εγώ θεωρώ ότι η Ρωσία είναι ένας εταίρος, είναι φυσικός ευρωπαϊκός χώρος αν θέλετε. Κύριε, ίσως πρόεδρε της Κομισιόν, αυτή η στήριξη σε μια κυβέρνηση που καταδίκασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πόσο θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ε, με την ε, κυβέρνηση της Ουκρανίας στην οποία συμμετέχουν ζει. Τι θα γίνει, θα μπούμε, θα συνεχίσουμε να είμαστε, να μας σέρνει το άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών. η Ρώσοι είναι εταίροι μας, δεν είναι εχθροί μας. Λίγο πολύ σας ανέφερα τα ερωτήματα. Από εκεί και πέρα φαντάζομαι θα εκλεγείτε αφού σας στηρίζουν και οι σοσιαλδημοκράτες, όμως εδώ έχετε έρθει ε, μπροστά στην αριστερή αντιπολίτευση. Υπάρχει και αυτό, τι να κάνουμε, δεν είναι όλοι υπέρ της Ευρώπης. Κύριε Γιούγκερ, δεν θα ε, πληρωθεί το χρέος Είστε ένας άνθρωπος ακέραιος. Ε, αν πάτε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα το δείτε ότι δεν μπορεί ο κόσμος να αποπληρώσει ε, και Έχουμε και την, ε, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που θέλουν να αλλάξουν το καταστατικό της. Μην καταστρέψουμε τα πάντα. Oh, merci Jean-Luc. Ευχαριστώ, Νεοκλής. Ε, <clears throat> είμαι ο Κλής ε, από την Κύπρο. Ε, κύριε Ιούγκερ, είστε ο υποψήφιος που προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Το κόμμα που κατά την άποψή μας ευθύνεται περισσότερο για τις νεοφιλεύθερες πολιτικές της σκληρής λιτότητας στην Ευρώπη. Υπήρξατε και πρόεδρος του Eurogroup που προώθησε αυτές τις πολιτικές. Το μνημονίο της Τρόικα που οδήγησαν ολόκληρες κοινωνίες ιδιαίτερα στον Νότο, στην εξαθλίωση, την αργία, τη φτωχοποίηση. Όντω αυτό που είπετε για το ΔΝΤ Ταμείο ισχύει. Η απάντηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι χρειαζόμαστε το Διεθνέ Νοματικό Ταμείο διότι έχει τεχνογνωσία. Ποια τεχνογνωσία έχει, νομίζω σήμερα τη βιώνουν οι λαοί τη Ευρώπη. Τη βιώσαν όμω για δεκαετίε οι χώρε του Νότιου ημισφαιρίου, οι αναπτυσσόμενε χώρε. Βίωσαν δηλαδή πολιτικέ λιτότητα, πολιτικές που διάλυσαν ολόκληρες χώρες και κοινωνίες. Το ερώτημα που προκύπτει όμως είναι δεν απαντήσατε, ενώ είπατε ότι είναι η θέση σας το ότι τι γύρευε το Διεθνή Ταμείο στην Ευρώπη, δεν απαντήσατε τι θα πράξετε σήμερα. Είπατε κάποια α, νεφολόδη α, ε, α, ε, ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Τρόικας, αλλά δεδομένης της προσήλωσης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στις νεοφιλεύθερες πολιτικής κληρινότητας, τι θα πράξετε ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη σχέση και τη συμμετοχή του Διεθνού Ματικού Ταμείου. Το δεύτερο ερώτημα που θέλω να σας ε, θέσω είναι για το Κυπριακό. Ε, τι θα κάνετε προκειμένου η Τουρκία να υλοποιήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις ως υποψήφια για ένταξη χώρα και να επιδείξει μια επικοδομητική στάση για την επίλυση του Κυπριακού. Η Κομισιόν έχει επαλημένα δηλώσει ότι θα στηρίξει τη διαδικασία των συνομιλιών για την επίτευξη λύσης. Τι είναι αυτό που θα πράξετε ώστε να βοηθήσετε αυτή τη διαδικασία για να φτάσουμε σε αίσιο πέρα σε αυτή τη διαδικασία και να επανενώσουμε την Κύπρο μας, αλλά και πώς ε, θα τοποθετηθείτε σε ενέργειες που, έχει, ε, που προωθούνται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και ιδιαίτερα μέτρα που προωθούνται για και εμβαθύνουν το χάσμα μεταξύ των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο. Οδηγούν δηλαδή σε μονιμοποίηση της κατοχής και της διέρεσης αντί να οδηγούν στην επανένωση. Και αναφέρομαι ιδιαίτερα σε αυτές τις προσπάθειες που καταβάλουν διάφοροι για προώθηση του απευθείας εμπορίου. Σας ευχαριστώ. Arvoisa Olen Merja Suomesta. από τη Φιλανδία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήλθατε κύριε Γιούγκερ. Η απογοήτευση του κόσμου σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων στην Ευρώπη και η αδύναμη δημοκρατική πρόοδος αποτυπώθηκε στο αποτέλεσμα των εκλογών γιατί ήταν σαφέ. Πώ θεωρείτε λοιπόν ότι θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτή την ανάγκη να προωθηθεί η δημοκρατία, η ανοχή στην Ευρώπη. Ευχαριστώ, Μέρια. Και τώρα, Άνια Χάζεγκαπ. Σας ευχαριστώ. Άνια Χάζεγκαμ από το κόμμα για τα ζώα στην Ολλανδία. Πρόκειται για ένα κόμμα το οποίο δεν ασχολείται μόνο με τα βραχυπρόθεσμα οικονομικά συμφέροντα για τον άνθρωπο, αλλά και για την προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος. Αναρωτιέμαι λοιπόν, ποιε είναι οι ιδέες σας για το τι μπορεί να βελτιωθεί εδώ στην Ευρώπη. Και έχω και κάποιες σύντομες ερωτήσεις να σας κάνω. Εδώ και χρόνια περιμένουμε ένα νόμο πλαίσιο για τα ζώα. Ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτίθεστε να φροντίσετε ο, νόμος αυτός να αποσταλεί το συντομότερο δυνατόν προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά δεύτερον, υπάρχουν πολλές, ε, παρανο... πολλά ακόμα ε, θέματα που μας απασχολούν στις διεθνείς μεταφορές ζώων που τα ε, κουβαλάνε από εδώ και από εκεί σε ακραίες καιρικές συνθήκες, σε μεγάλα κρύα, σε μεγάλους καύσονες. Είστε διατεθειμένος ε, να πιέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση της ε, οδηγίας για τις μεταφορές των ζώων. Και τέλος, μία ερώτηση για την ε, συνθήκη της Λισαβόνας, όπου αναφέρεται ότι τα ζώα έχουν και αισθήματα και ότι θα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη. Αλλά γίνεται εξαίρεση για θρησκευτικούς και πολιτισμικούς σκοπούς, στις οποίες περιπτώσεις επιτρέπονται ακραίες φρικαλαιότητες κατά των ζώων, όπως για παράδειγμα οι ταυρομαχίες στην Πορτογαλία, στην Κύπρο, την Πορτογαλία, την ε, Μάλτα, κυνήγι άγριων πτηνών. Εγώ μπορώ να συνεχίσω ε, επί ώρες βάρβαρες πρακτικές, ε, οι οποίες δεν μπορούν να διατηρηθούν Προβλέπετε λοιπόν τέτοιες δυνατότητες ε, προκειμένου αυτές οι βιαιότητες, αυτές οι φρικαλαιότητες να περιοριστούν και να καταργηθούν. Και τέλος πιστεύω ότι οι αγροτικές επιτετήσεις θα πρέπει να καταργηθούν και θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος αυτό το γύρο είναι ο Γιώργος Ζουτράν αλλά να πω ότι θα προσθέσουμε δύο ομιλητές σε αυτό το γύρο, προκειμένου όλες οι αντιπροσωπείες να έχουν το δυνατότητα να μιλήσουν. Γιώζου και με Λουκ, Λουκ Πλάνεγκαν και μετά η Μαρίζα Ματίας. Γιώζου, πείτε. Ευχαριστώ, Γκάμπ. Καλημέρα σας. Ε, λέγομαι Γιώσου Αρίστη. Είμαι Βάσκος. Δύο πολύ σύντομα ερωτήματα. Η κοινωνική πλειοψηφία τη χώρα των Βάσκων στηρίζει την ερηνευτική διαδικασία και θα πρέπει και το κράτος, ε, το Ισπανικό, να κάνει κάποια βήματα στη διαδικασία. Δεν το κάνει. Εσείς, σας ερωτώ, ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα στηρίξετε το αίτημα της πλειοψηφίας της κοινωνίας, ε, θα ε, προωθήσετε την ανάπτυξη της ειρηνευτικής διαδικασίας. Και φυσικά και εμείς θα είμαστε στη διάθεσή σας να σας δώσουμε κάθε πληροφορία για να απαντήσουμε σε όλα σας τα ερωτήματα. Δεύτερο ερώτημα. Η ομάδα του Μπαρόσο απέναντι στο καταλανικό και σκοτσέζικο δημοψήφισμα και το μέλλον των ε, δύο λαών ε, επηρεάστηκε πάρα πολύ από αυτά που λένε οι κυβερνήσεις. Ε, εσείς τι πιστεύετε, μπορούν να αποφασίζουν ελεύθερα οι Καταλανοί, οι Σκοτσέζοι και οι Βάσκοι αύριο μπορούν να έχουν αυτό το δικαίωμα να αποφασίσουν ελεύθερα. Ευχαριστώ γιος. Ο Λουκ έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε. Καταρχάς, να μην μπλέκετε την Ευρώπη, νομίζω, την Ευρώπη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ λατρεύω, αγαπώ την Ευρώπη, αλλά απεχτάνομαι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ξέρετε, ε, η Ιρλανδία 67 δισεκατομμύρια ευρώ έχει τέτοια και 42% της διάστασης για 1% του πληθυσμού. Εμείς θέλουμε λοιπόν πίσω τα χρήματά μας. Στις 31 Μαΐου του 2012 έκαναμε δημοψήφισμα για το ESA και τι αποφασίστηκε αναδρομικά να έχουμε επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Να πάρουμε τα λεφτά μας πίσω δηλαδή. Σήμερα είμαστε στο 1,2-3 ε, δισεκατομμύρια που έχουμε δώσει σε αυτό το σύστημα. Λίγο, λίγο λοιπόν μας ε, ε, ταΐζουν ψέματα οι κυβερνήσεις μας. Ε, στο 2012 ε, τον Ιούνιο ε, περιγράφηκε μία αλλαγή στην ευρωπαϊκή πολιτική σε ό,τι αφορά την αναδρομική επανακεφαλοποίηση των τραπεζών και μας είπαν ότι θα μας έδιναν πίσω τα χρήματά μας. Τον Οκτώβριο του 2012 διεθνώς αναφέρθηκε ότι η Ιρλανδία ήταν η ειδική περίπτωση και ότι η καγκελάριος Μέρκελ μαζί με τον δικό μας τον ηγέτη συνήλθαν και αποφάσισαν ότι είμαστε ιδιαίτεροι περίπτωση. Ιανουάριο του 2013, ο Υπουργό Οικονομικών μα μας είπε ότι η Γερμανία και η Γαλλία μα φιλούσαν. Γιατί μα φιλούσαν δηλαδή, να μα καρφώσουν πίσω όπλατα, έτσι φαίνεται. Στην 2014, Γενάρη, μα είπατε ότι ξέρουμε τι εκπροσωπούμε. Εσεί ξέρετε τι εκπροσωπείτε. Για την Ιρλανδία είπατε ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο βαθμό αναδρομικότητα στο μηχανισμό, εντάλλως θα χάσει κάθε νόημα. Και αυτό φαίνεται λοιπόν ότι ήταν ένα ψέμα για την διαδικασία υποψηφιότητά σας, για να πείσετε τον κόσμο να ψηφίσει το ΕΛΚ. Γιατί από τις εκλογές και μετά μας λένε τώρα τι μας λένε, ότι δεν θα πάρουμε πίσω τα χρήματά μας. Τρεις υποψήφοι λοιπόν από την Ιρλανδία, τρεις ε, βουλευτές από το Φινιγκέιλε ε, κλέχθηκαν και βάσει ψεμάτων σα ψήφισαν, σα υποστηρίξαν. Ρωτώ λοιπόν γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει να ζητά τέτοιο ε, βαρύ φορτίο από την Ιρλανδία και ο, τα δισεκατομμύρια τα οποία χρειάστηκαν για να σωθούν ε, τράπεζε ζόμπι και για την Ιρλανδία και για όλη την Ευρώπη. Δεν έχει θυσιάσει αρκετά πια η Ιρλανδία. Εμείς θέλαμε μια κοινότητα, μια κοινότητα δεν ε, παίρνει το ψωμί από το στόμα του κόσμου για να ταΐσει τις τράπεζες. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά, μεγάλα ηγέτη του μέλλοντος. Okay. Danke, Luke. Μάλιστα, Λουκ. Ευχαριστώ. Μαρία Ζαματίας. Ε, Μαρίζα Ματίας από τον μπλόκο τη Κέρδα, Πορτογαλία. Ε, κύριε Γιούνκερ, γνωριζόμαστε γιατί έχουν γίνει πάρα πολλέ ακροάσεις στην ΕΚΟΝ ε, όπου παρευρεθήκαμε και οι δύο ξέρουμε, τα έχουμε πει για τι πολιτικές λιτότητε, για την πολιτική της Τρόικα ε, και περνάω τώρα σε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, ήσασταν ε, Πρωθυπουργό σε μια χώρα όπου ανθεί η κερδοσκοπία στην Ευρώπη ε, και Ταυτόχρονα είσαστε από τους λίγους ε, στις ακροάσεις ΕΚΟΝ που κατέκριναν τις πολιτικές λιτότητες. Οπότε ποιο να πιστέψουμε, τι, τι, ποιο από τα δύο θα υποστηρίξετε αν γίνετε πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεύτερον, για το χρέος. Ε, δεν με απαντήσατε για την αναδιάρθρωση του χρέους. Ε, κάθε φορά που υπάρχει συνένεση στις χώρες του Νότου για την αναδιάρθρωση του χρέους, διότι πρόκειται για μια κρίση δημοσίου χρέους και όχι πλέον μια χρηματοοικονομική κρίση και οι φτωχοί πληρώνουν την κρίση που δεν προκάλεσαν. Ε, πώς θα γίνει βιώσιμο το χρέος. Ε, δεν θα σταματήσει πουθενά αυτό. Εάν δεν αναδιαρθρωθεί το χρέος ποτέ δεν θα γίνει βιώσιμο. Πώς τοποθετήσετε γι' αυτό. Τρίτη ερώτηση ε, για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Πολύ σύντομα. Τι θα κάνετε για τις ε, χώρες ε, που δεν ε, θα τηρούν το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, γιατί είναι αδύνατον να το τηρήσει κανείς και ξέρετε ότι δεν θα το τηρήσουν οι χώρες. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αποτελειώσει τις χώρες ή θα αποτελειώσει επιτέλους το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Και τελευταία ερώτηση πραγματικά για τη μετανάστευση. Μιλήσατε για νόμιμη και παράνομη μετανάστευση, πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, τέλος πάντων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Ευρωπαϊκό χώρο Μιλάμε για ε, παράνομη μετανάστες που ε, κατά παραβίαση της συνθήκης. Ε, άρα δεν ισχύει η ελεύθερη μετακίνηση των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πολίτες που 20-30 χρόνια δουλεύουν σε ένα κράτος μέλος και τους επαναπροωθούν στις χώρες τους. Δεν είναι απαράδεκτο αυτό είναι πολύ ελαστική νόμη για την αγορά εργασίας και πάρα πολύ αυστηρή, αυστηρή για την μετανάστευση. Τι πρόκειται να κάνει γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πρωτού σας δώσω το λόγο. Θα, κύριε Γιούγκερ, θα ήθελα να πω ότι έχουμε ακούσει από τις αντιπροσωπείες όλο το εύρος των αντιπροσωπιών. Και έχω δέκα ε, άτομα που ζητούν το λόγο, τουλάχιστον στη λίστα. Και θα προτείνω ότι να κλείσουμε μετά. Να δώσουμε τη δυνατότητα στον κύριο Γιούνκερ να απαντήσει στις ερωτήσεις που προέκυψαν τώρα. Και έχουν να κάνουν ουσιαστικά με την δομή του χρέους, με την πολιτική αυτή. Πώς θα συνεχιστεί, πώς πρέπει να συνεχιστεί η πολιτική σε ό,τι αφορά. Και να περάσουμε στο θέμα της μετανάστευσης. Κυρίως αυτό το κομμάτι είναι εκρεμές, είναι ασαφές. Πώς μπορεί λοιπόν ε, να ασκηθεί μια διαφορετική πολιτική για τη μετανάστευση, προκειμένου να υπάρχει νόμιμη μετανάστευση, νόμιμη πολιτική ασύλου. Πώς αυτό μπορεί να αλλάξει και την πολιτική στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ό,τι αφορά ε, το φορτίο στα εξωτερικά σύνορα. Δεν θα πρέπει να υπερβούμε τα 10 λεπτά γιατί στην περίπτωση αυτή οι διερμηνείς ε, που πραγματικά ήδη εργάζονται πέρα από το ωράριό τους ε, θα πρέπει να φύγουν. Κύριε Πρόεδρε, το ίδιο και εγώ, το ίδιο και εγώ όπως και κυρία Πέδρε. Γιατί έπρεπε να έχουμε ολοκληρώσει πριν από ένα τέταρτο, αλλά δεν έχουμε ολοκληρώσει και, ε, και εγώ θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτό το ευρωπαϊκό ωράριο, γιατί θα ήθελα τουλάχιστον 5 λεπτά. Ώρα να παυσίσει. Ε, θέλω να επανέλθω σε κάποια ερωτήματα, ήταν πολύ άριθμα. Πρώτα απ' όλα, για την TTIP, το Διατλαντικό Σύμφωνο με τη ΣΥΠΑ, που με ενδιαφέρει και με ανησυχεί. Η Ευρώπη για κάποιες αρχές δεν μπορεί να αλλάξει ε, επειδή έτσι το θέλουν οι Αμερικάνοι ε, το εργατικό δίκαιο, τους κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ούτω καθεξής. Ε, στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων δεν θα γίνει αυτό για την προστασία των δεδομένων όλος ιδιαίτερος πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι δεν θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης αυτό το ζήτημα. Ε, υπάρχει η εξή αρχή ότι όσοι ε, έχουν εμπορικέ διαπραγματεύσει εδώ στην Ευρώπη και η επιχείρησή τους έχει την έδρα τη ε, στην Ευρώπη πρέπει να συμμορφώνεται με το δικό μας δίκαιο. Δεν είμαστε θα υπερασπιστούμε αυτές τις αξίες και δεν πρόκειται να επέλθει καμία αλλαγή. Θα πρέπει ε, να αναλογιστούμε ε, και να εξετάσουμε προσεκτικά τα μελλοντικά ε, βήματα. Τώρα το Λουξεμβούργο σε κανένα μαύρο κατάλληλο δεν είναι κανενός διεθνούς οργανισμού. Θυμηθείτε και πέρσι στον κατάλογο του ΟΣΑ δεν είμαστε σε καμία μαύρη λίστα. Ε, κύριε Μελανσόν, όταν ε, μιλάτε για τη Ρουσία, ε, παρότι θα συμφωνήσω εν μέρη με την ανάλυση σας για τις Ουκρανικές αρχές, πρέπει να δεχτούμε το προφανές ότι η Ρωσία είναι πολύ σημαντικός εταίρος και παραμένει ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, το χαρτί της ασφάλειας ε, αφορά και τον συναρχιτέκτον αν θέλετε του εγχειρήματος της ασφάλειας που είναι η Ρωσία όσοι δεν με ψήφισαν, ψήφισαν για την πρότασή μου στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησαν ε, ε, μαζί μου για το πώς βλέπω τη Ρωσία. Εγώ πιστεύω ότι ε, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αμφισβητήσουμε τη στρατηγική σημασία της εταιρική σχέσης μας με τη Ρωσία και φυσικά όταν παραβιάζονται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να το συζητάμε ανοιχτά αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη Ρωσία όπως στην εποχή του ψυχρού πολέμου. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προσυπογράψω αυτά. Που λέτε, για την Κύπρο. Κοιτάξτε, είναι μία διαδικασία που γίνεται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Δεν ε, έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή η διαδικασία μπορεί κανείς ε, ε, να το επιθυμήσει. Αφήνουμε το θέμα στα χέρια ενός άλλου διεθνούς οργανισμού αυτό το ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα κομμάτι των εργασιών συμμετέχει αλλά δεν έχει μια συνολική εικόνα. Μίλησα με πολλούς Κυπρίους φίλους για να βρούμε τρόπους ε, με τους οποίους θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε στη διαπραγματευτική δομή το ρόλο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εύκολο δεν είναι. Ναι, για το δίκαιο των ζώων. Ε, είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να έχουν νομοθεσία για το ευσύν των ζώων. Είναι ζώντες οργανισμοί και δεν είναι αντικείμενα υπάρχουν πολυάριθμες ε, συμβάσεις ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη μεταφορά των ζώων και για άλλα ε, ζητήματα στα οποία αναφερθήκατε κυρία μου και είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος μιλάμε για αυτά τα ζητήματα, γιατί είμαι και στο ε, Διεθνές Συμβούλιο της Λίγας Προστασίας των Ζών για να ξέρετε ε, σε ποιον απευθύνεστε. Ε, δεν, ποτέ δεν ήμουν σε κάποια επιχείρηση, αλλά έδινα νομικές συμβουλές μέχρι πρότινος στην Διεθνή Λίγα Προστασίας των Ζών για να ξέρετε. Ε, ζητώ συγγνώμη που το λέω, αλλά με ρωτάνε, κυρία Βαζιά, ε, εκτός μικροφώνου, κυρία Βαζιά λέει για αναφέρεται σε αυτό που είπε ο κύριος Γιούνκερ ότι ήταν ε, νομικός σύμβουλος για τη Λίγα προστασία των Ζώων. <clears throat> Κοιτάξτε, ναι, τώρα δεν είμαι, εν πάση περιπτώσει. Έκανα λάθος το χρόνο. Τώρα δεν είμαι νομικό σύμβουλο. Ε, αποχώρησα. Ε, ε, ξέρετε τώρα για τα θέματα ανεξαρτησίας σέβομαι ε, τη συνταγματική τάξη και την κυριαρχία των κρατών μελών ε, δεν μπορώ να παρέμβω σε αυτή τη συζήτηση που ε, άπτεται της, της εθνικής κυριαρχίας, ε, σέβομαι τη συνταγματική τάξη των κρατών μελών, πρέπει ε, τις αποφάσεις ε, της συνταγματικής ε, δικαιοδοσίας να τις σεβόμαστε. Ξέρω πού μπορεί να οδηγήσουν αυτά τα δημοψηφίσματα η ε, οποία θα ε, τηρήσω ε, για αυτό το ζήτημα. Για το Σύμφωνο Σταθερότητας θα σας πω ότι θα εφαρμοστεί ως έχει με λογικό τρόπο και έχοντας και μία κλίδα ανάγνωσης πιο οικονομικού χαρακτήρα. Τώρα για την ε, μηχανή λιτότητας ε, του ΕΛ και τα λοιπά. Κοιτάξτε, θα σας πω ένα πράγμα. Η νεοφιλελεύθερη, η, πολι... η φιλελεύθερη πολιτική και το νεοφιλελεύθερο κομμάτι είναι έργα του κυρίου Μπλερ και του κυρίου Σρέντερ. Εγώ ποτέ δεν θα ε, είχα εγκρίνει μια τέτοια νομοθεσία γιατί πάντοτε αγωνιζόμουν για την απορρίθμιση μπορείτε να μιλείτε συντηρητικό, μπορείτε... Εκτός μικροφώνου ο κύριος Μελανσόν, τέλος πάντων έχω γνωρίσει οι αριστερές κυβερνήσεις όπου τα καλύτερα μέλη της ε, ακολουθούσαν πολύ διαφορετική πορεία και επίσης έχω συνεργαστεί με τέτοιες κυβερνήσεις και ξέρω ποιος ακριβώς ευθύνεται για τις φιλελεύθερες πολιτικές στην Ευρώπη δεν ευθύνομαι εγώ ε, ο κύριος Μελανσόν και εγώ ίδιος πεινάμε, οπότε πρέπει να αποχωρήσουμε. Ευχαριστώ, ήταν πολύ ευχάριστη συζήτηση μαζί σας. Σας ευχαριστούμε και πάλι.